Τεύματα πολιτών, ομάδων ε, πολιτών και οργανώσεων για την προαγωγή καλύτερη συνεννόηση και συμφιλίωση με στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δραστηριότητε που αποτελούν συγκεκριμένη έκφραση των αξιών που καταγράφονται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι βραβευθέντε δραστηριοποιούνται σε πολύ διαφορετικού τομεί, όπω ο διαπολιτισμικό διάλογο, η αλληλεγγύη, η ισότητα, η κοινωνική ενσωμάτωση, η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης. Στις 5 το απόγευμα σήμερα θα γίνει μια πανηγυρική παρουσίαση των των αυτών πολιτών. Σας καλούμε όλους και βεβαίως σήμερα έχουμε εδώ μέσα στην γαλαρία ε, ε, τους πολίτες αυτούς, μερικούς από τους πολίτες αυτούς, οποίους και χαιρετίζουμε.